<laughs> Ξεκινάει η συνεδρίασή μας. Θα εξετάσουμε τώρα τη δήλωση της Επιτροπής Διαρθρώσεις υποδοχή για τα Παιδιά Στόχη της Βαρκελόνης. Το λόγο έχει ο Επίτροπος Σπίτλα. Καλώς ήρθατε κύριε Σπίτλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.